σχετικά με ζητήματα λία στο πλαίσιο τη Διεθνού Συμφωνία για τη θαλάσσια βιοπικιλότητα σε περιοχέ που βρίσκονται εκτό εθνική δικαιοδοσία. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστώσω τους Σκιώδης για την πολύ καλή συνεργασία κατά την επεξεργασία αυτής της έκθεσης. Η έκθεση αυτή αποστέλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ως ε, υποστήριξη προς την Επιτροπή και ξεκαθαρίζει τις προτεραιότητες της δικής μας Επιτροπής όσον αφορά μια νέα σύμβαση. Ως γνωστόν, 65% των θαλασσών ε, δεν καλύπτονται από το δίκαιο της θάλασσας. Πρόκειται λοιπόν για μια βιώσιμη διαχείριση εδώ ε, θαλάσσιων περιοχών που δεν ε, καλύπτονται μέχρι στιγμής. Γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει και ψάχνουμε τρόφιμα εν ώψη και της αύξησης του πληθυσμού της ε, γης. Και μελλοντικά θα πρέπει όλες αυτές οι προσπάθειες να επικυρωθούν και να προσαρμοστούν στην, στις νέες πραγματικότητες. Ε, σημαντική συμφωνία είναι αυτή που αφορά τα ηχθειοαποθέματα. Ε, υπάρχει μια συμφωνία από το 1995 που αφορά ορισμένα μετανασταυτικά είδη και βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν τη σύμβαση αυτή. Η Επιτροπή είναι ωστόσο υπέρ της διατήρησης αυτών των μέτρων και στο πλαίσιο ενός ε, μελλοντικού εξυγχρονισμού. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ε, έχει αποφασίσει ότι ε, θα πρέπει να γίνουν κάποιες διαπραγματεύσεις και το 2015 συστάθηκε μια άτυπη ομάδα εργασίας ad hoc. Ελπίζουμε λοιπόν ότι σύντομα θα έχουμε μια νέα έκθεση. Η Επιτροπή μας ε, προσπαθεί να εργαστεί για την εκπόνηση, συγγνώμη, ενός νομικά δεσμευτικού πλαισίου όσον αφορά τη σύναψη μιας ε, νέας ε, σύμβασης. Η Επιτροπή ήταν ιδιαίτερος καθοριστική, ο ρόλος της Επιτροπής αντιτέλους καθοριστικός για αυτή τη σύμβαση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες ξερούνται από αυτή τη σύμβαση, από αυτές τις συμφωνίες ε, και θεωρείται ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να ρυθμίζονται εθνικά. Ωστόσο, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε η Κομισιόν είναι σύμφωνη με αυτές τις ε, εξαιρέσεις. Αυτό λοιπόν για μας συνιστά μια προτεραιότητα. Αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να δεχτεί μέσα μια παραδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας του 95 όσον αφορά τα αποθέματα. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα συμπεριληφθεί στη νέα συμφωνία. Επίσης θα πρέπει να αυξηθεί η σημασία του νέου οργανισμού για τη διαχείριση της αλίας. Γιατί οι δραστηριότητες του οργανισμού αυτού ήταν ιδιαίτερως θετικές όσο και των περιφερειακών οργανώσεων για τη διαχείριση της αλίας. Ε, θα πρέπει όλες οι χώρες να συμμετάσχουν σε αυτούς τους οργανισμούς παράκτη λέει δεν μπορεί να τελεσφορήσει παρά μόνο αν υπάρχει ένας επαρκής συντανισμός όλων των δραστηριοτήτων. Και ε, θα πρέπει βεβαίω να υπάρξει και μία ε, εξασφαλισμένη προστασία της ε, βιοπικιλότητας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Γκαμπριέλ Μάτο για ένα λεπτό. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συγχαρητήρια πρώτα πρώτα προ τον εισηγητή. Θέλω να σα πω ότι αυτό το οποίο συζητήσαμε ε, πρόκειται για ένα ε, όργανο του διεθνού δικαίου, συμφωνία διεθνού δικαίου για να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε, αλλά δεν χρειαζόμαστε υπέρ τη νομοθεσία, διότι το υπάρχον πλαίσιο είναι επαρκέ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι όλοι οι συμβαλόμενοι να τηρούν τα συμπεφωνημένα διότι έτσι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Μέχρι σήμερα είναι προφανές ότι δεν τα πήγαμε και τόσο καλά, γιατί δεν είμαστε αποτελεσματικοί όσον αφορά τη χρήση ε, του πλαισίου που υπάρχει και οι περιφερειακές αρχές αλληλείας έχουν την αρμοδιότητα. Θα πρέπει να διαχειριστούν τους αλληλευτικούς πόρους, θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους όπως και σήμερα. επομένω θα πρέπει εμείς να αναβαθμίσουμε, θα πρέπει να ενισχύσουμε τον συντονισμό μεταξύ των διεθνών οργανισμών και περιφερειακών οργανισμών και θα πρέπει να εργαστούν συντονισμένα και έτσι να προστατεύσουν τους παγκόσμιους διευθυντικούς πόρους αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σάντος είναι επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τον εισηγητή. Κύριε Επίτροπε, η ΑΕΛΗ έχει να κάνει με την βιοπικιλότητα και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, επιβίωση των κοινοτήτων των ε, αλλιέων αλλά χρειάζεται να γίνει μια προσέγγιση επιστημονική να λάβουμε υπόψη τα οικοσυστήματα και τα EBSAs θα πρέπει ομένως να δούμε ότι θα πρέπει να προστατευτούν οι ελευθερικοί πόροι και θα πρέπει να προστατεύσουμε και την βιοπικιλότητα. Αυτά και είναι τον κόσμο. Άρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την έκθεση στην προσέγγιση που υιοθετεί και έτσι να προστατευτούν οι θάλασσες και οι ωκεανοί εκτός εθνικής διοικειοδοσίας.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 συγκεκριμένα τονίστηκε ότι πρέπει να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος και έτσι θα πρέπει η αλλιευτική βιομηχανία και η αγορά της ευρωπαϊκής ένωσης να είναι προσανατολισμένες προς την βιωσιμότητα. η σύμβαση αυτή του οηε πρέπει να εφαρμοστεί βεβαίως από όλες τις χώρες όχι μόνο τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και τις χώρες οι οποίες είναι υποψήφιες προς ένταξη στην ευρωπαϊκή ένωση και τις υπόλοιπες ταυτόχρονα εκτός από την προστασία των πόρων νομίζω ότι θα πρέπει για άλλη μια φορά να επισημάνω ότι η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει επιτέλους να ασχοληθεί σοβαρά για την στήριξη των αλλιέων όλων των κρατών μελών και ιδίως της πατρίδας μου της ελλάδος. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η διατήρηση της ε, βιοπικιλότητας ε, προποθέτει έναν καλό συντονισμό και μια συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι το πιο ενδεδειγμένο φόρουμ προκειμένου να να ενισχυθούν οι προσπάθειες ε, συνεργασίας και συντονισμού για την καλή διατήρηση των ηχθειοποθεμάτων. Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι το δεδειγμένο εργαλείο προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμαστούν θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές γνώσεις και σωστή αξιολόγηση του αντικτύπου των ελευτικών δραστηριοτήτων. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα να δερματίσει ένα καθοριστικό ρόλο ε, στο πλαίσιο της αλληλευτικής ε, πολιτικής. Ο κύριος Πόλτσακ έχει το λόγο. Θα ήθελα να υποστηρίξω όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στο θέμα της αποψινής μας ε, συζήτησης δηλαδή σε μια βιώσιμη εξέλιξη των θαλασσών, της αλίας και της ε, βιοπικιλότητας των θαλασσών. Από την άλλη θα πρέπει να μας είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με εξελίξεις που έχουν σαν, που είναι εις βάρος της ε, βιοπικιλότητας. Για παράδειγμα το γεγονός ότι παράκτες ε, περιοχές αστικοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Ακόμα και η εντατικότητα της ε, αλίας, η οποία βεβαίως απειλεί την επιβίωση των ηχθειοαποθεμάτων. αποθεμάτων καθώς και η ρήπανση των υδάτων ε, λόγω των αληφτικών ε, στόλων. Χαιρετίζω βεβαίως την έκθεση αυτή. Ο κύριος Καπούτο έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Τη σωστή στιγμή, αλλά και ίσως με λίγο καθυστέρηση ήρθε αυτό το νομοθέτημα, τόσο ώστε να προστατεύσουμε η βιοποικιλότητα στις περιοχές εκλήγει για αύξηση των δικαιοδοσιών και τώρα επομένως ε, επεβάλλεται να φροντίσουμε για τους αληθικούς πόρους χωρίς άλλη καθυστέρηση χρειάζεται να υπάρξει ε, μια σύμβαση ε, για το δίκαιο της θάλασσας η οποία να είναι δεσμευτική και θα πρέπει να καλυφθεί πάσα λεπτή δραστηριότητα και γι' αυτό έχουμε τώρα αυτήν την σύμβαση και θα πρέπει να αναγνωριστεί η σημασία της οικολογίας για την ε, θάλασσα. Έχουμε αυτήν την ε, νέα σύμβαση. Προβλέπει το να υπάρξει ένα όργανο διεθνού δικαίου για να προστατεύσει το περιβάλλον για κάποιες δραστηριότητε που μπορούν να έχουν κάποιες επιπτώσεις σημαντικές ε, για τις θάλασσες και τους ωκεανούς οπότε χρειάζεται να προστατεύσουμε και το περιβάλλον αλλά και να έχουμε μια κοινωνική και οικονομική πολιτική. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ξέχασα τον κύριο Κούν και επειδή έχουμε κάποιο χρόνο, έχετε το λόγο κύριε Κούν. Ε, κυρία Πρόεδρε, μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις όπου ακούγονται πολλές ε, διαφορετικές ε, απόψεις και όπου κανείς μπορεί να προβάλλει κάποια επιχειρήματα η εφαρμογή αυτής της διεθνούς σύμβασης ε, είναι το ζητούμενο γιατί υπάρχουν τα αντίστοιχα νομοθετήματα όπως είπε και ο κύριος Μάτο αλλά θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχυθούμε όσον αφορά τη θέση μας στην αγορά 70% ε, των διαφόρων ε, των ψαριών και των προϊόντων από ψάρια είναι εισαγωγές και ένα μεγάλο ποσοστό προέρχονται από ηχθειοκαλλιέργειες. Ε, οι Ασιάτες ε, και άλλοι εξάγουν στην Ευρώπη και γι' αυτό θα πρέπει το κοινό αίτημα να είναι ε, ένα κοινό eco-label το οποίο θα πρέπει να είναι στα προπόθεση για αυτές τις αγωγές, αλλιώς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκές αγορές. Και τώρα ο κύριος Βέλλας έχει το λόγο εξ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Καταρχήν θέλω να πω ότι η έκθεση ιδίες πρωτοβουλίας για την ε, αλληλεία είναι ευπρόσδεκτη. Η έκθεση αφορά την ε, ε, βιώσιμη χρήση των της βιοποικιλότητας ε, σε περιοχές ε, εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Είναι σημαντικό που δίνουμε έμφαση σε αυτή τη σημαντική εξέλιξη που πρέπει να ε, φέρει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας σε ευθεία γραμμή με τις πρόσφατες εξελίξεις. Η έκθεση αυτή της κυρίας Νικολάη, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, έρχεται την κατάλληλη στιγμή ως δεδομένο ότι η πρώτη Παρασκευαστική Επιτροπή που ξεκινά τις διαπραγματεύσεις έχει μόλις συνεδριάσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες μεταξύ της 28 Μαρτίου έως της 8 Απριλίου θα ακολουθήσει μια δεύτερη συνεδρίαση στο τέλος Αυγούστου μεταξύ 26 και Αυγούστου και 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση σωστά επισημαίνει ότι το νέο νομικό μέσο θα ασχοληθεί με διάφορα στοιχεία όπως η θαλάσσια γενετική πόρη συμπεριλαμβανομένου και του θέματος της κατανομής των ωφελών, το θέμα των ε, της διαχείρισης, εργαλείων διαχείρισης και των προστατευόμενων περιοχών και την ε, τεχνολογία της θάλασσας. Ένας από τους βασικούς στόχους της νέας αυτής συμφωνίας είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα επιτρέψει τη δημιουργία και τη διαχείριση των θαλασσίων προστατευόμενων περιοχών έτσι ώστε θα να μπορέσει η παγκόσμια η, κοινότητα να τηρήσει το στόχο της διάσκεψης του Ρίο για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη ότι το 10% θα πρέπει να έχει επιτευχθεί μέχρι το 2020. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ε, λάβει υπόψη του τις, ε, και να εφαρμόσει τις διατάξεις της ε, UNCLOS, της σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, στην πράξη που αφορούν και την θαλάσσια βιοπικιλότητα. Όλα αυτά στην ανοιχτή θάλασσα μπορούν να επηρεάσουν, που μπορούν να επηρεάσουν την βιοπικιλότητα ποιότητα της θάλασσας πρέπει να ληφθούν υπόψη στη νέα συμφωνία χωρίς όμως να ε, υπονομεύσουν την, ε, τον, το, τον νόμο για το δίκαιο της θάλασσας. Συμφωνούμε με την έκθεση ότι το UNFSA συνεχίζει να λειτουργεί καλά και δεν θα πρέπει να ανοίξει και πάλι αλλά να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί καλύτερα. Εξακολουθούμε να στηρίζουμε ε, την εργασία των ΠΟΔΕ και πρέπει, θέλω να εξασφαλίσω ότι θα γίνουν πιο αποδοτικοί στην ε, διαχείριση των ε, εξαιρετικά μεταναστευτικών αποθεμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παίζει ε, κυρίαρχο ρόλο στις διαπραγματεύσεις και να υπερασπίζεται την ανάγκη προστασίας της θαλάσσιας βιοπικιλότητας σύμφωνα με τις διεθνείς μας διεσμεύσεις. Επίσης θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την, ε, ε, τις εργασίες των για τη διαχείριση της αλίας. Πρέπει να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην διατήρηση και την βιώσιμη χρήση, όπως έχει γίνει και με την πιο πρόσφατη CFP. Επίσης, δεν θα επιτρέψουμε στις διαπραγματεύσεις αυτές να διαταράξουν την ισορροπία των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων ε, που επιτεύχθηκε για ε, στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας γιατί σύμφωνα με αυτή όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να, μπορούν να αναλυφθούν. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την υποστήριξή σας ε, στην, στον αγώνα μας κατά της αδήλωτης παράνομη και παράνομης αλληλείας και προς, είναι ένα σοβαρό ε, ε, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόβλημα. Σας ευχαριστώ θερμά. The debate is closed. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο κύριο Βέλα.